Okay, friends. Uh, then we start. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ας ε, συνεχίσουμε με το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Θα δώσω το λόγο στην συγκήτρια Μαρία Αρένα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα η πρόταση της Κομισιόν είναι ενδιαφέρουσα. Την έχουμε εμπλουτίσει με διάφορα στοιχεία όπως τη συμπεριλήψη στατιστικών στοιχείων για την ποιότητα της απασχόλησης, και την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης αναπτύξη των ΗΕ, ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης επί της ευρωπαϊκής αγοράς, τον καθορισμό της ανάπτυξης και της παραγωγής βάσει άλλων κριτηρίων πέραν του απλού εγχώριου ε, καθαρού προϊόντος, ε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πτυχή της ισότητας των ανθρώπων στο πλαίσιο του στατιστικού προγράμματος. Εγώ έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες που κατατάσσονται σε τέσσερις συμβιβασμούς για τα θέματα ως εξή ε, τις ε, ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες, τη δημογραφική εξέλιξη, επισημένοντας τις επιπτώσεις της αστικοποίησης, καθώς και τη δυνατότητα των περιοχών αραιού πληθυσμού να παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι δύσκολο λόγω του μικρότερου πληθυσμού. Εκεί έχουμε υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. Δεύτερο συμβιβασμό για του πιο ευάλωτου ανθρώπου, τους αστέγους, ε, τους αναπήρους ή τις μειονότητες. Ε, Τρίτο συμβαστική δείκτες απασχόλησης και ανεργίας στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης και μετά η σύνδεση μεταξύ παραγωγικότητας και απασχόλησης καθώς και η χρήση δικτών που επιτρέπουν να δούμε πώς εξελίσσονται οι οικονομικές ανισότητες και η φτώχεια. Πιστεύω ότι αυτά τα τέσσερα θέματα θα μας βοηθήσουν να κατατάξουμε τις περισσότερες τροπολογίες που προτάθηκαν ε, και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ε, καθισχάσουμε τις ανησυχίε των ομάδων που υπέβαλαν τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνουμε τώρα το λόγο στους εισηγητές. Ε, κυρία Λόπεθ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ είμαι πεπισμένος ότι ε, υπάρχει μια αδρία συνέντευξη μεταξύ μας. Την Πέμπτη θα συναντηθούν οι σκιώδεις και εγώ επίσης συμφωνώ με πολλές από τις τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μερικές διαφοροποίησεις, να κρατήσουμε τις κύριες γραμμές της πρότασης Κομισιόν. Η πρόταση αυτή για μένα είναι μια θετική πρόταση και το στατιστικό πρόγραμμα της Κομισιόν θα υποστηρίξει τις προτεραιότητες της Κομισιόν εν ώψη του 2020. Αυτό το οποίο δεν συμφωνώ είναι η συμπερίληψη των 17 στόχων των Ηνωμένων για την Ανάπτυξη. Προφανώς είναι σημαντική η στόχη αυτή, αλλά δεν βλέπω πολύ καλά πώς συνδέονται με αυτό το θέμα που μας απασχολεί, πώς εμπλέκονται σε αυτό το στατιστικό πρόγραμμα, κατά τα άλλα που φαίνεται ότι όλα αυτά που είπε η συγήτρια κυρία Ρένα είναι πολύ θετικά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική συνένεση μεταξύ μας, μπορεί να υπάρξουν κάποια σημεία όπου θα υπάρξουν διαφοροποίησεις, θα είναι φυσικά καλό για όλους μας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ μας ως εισηγητές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκυρίκ από το ECR δεν είναι εδώ. Ούτε τον αντικαθιστά κανείς. Άλντε. Ο κύριος Σαμπόν δεν είναι εδώ. Είναι κανείς που τον αντικαθιστά. Κυρία Χάρκιν, όχι. Κύριε Σελίμωβιτς, όχι. Καλά. Κούε. Δεν είναι κανείς εδώ να εκπροσωπήσει την Κούε. Πράσινη. Τους εκπροσωπείτε εσείς. Όχι. Η κυρία Ζανόκα δεν είναι εδώ. Κύριε Μαρτά. Ούτε εσείς. Άρα μπορούμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Βάρερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δουλεύω στη Eurostat, είμαι διευθυντής και χαίρομαι πολύ που θα σας πω ορισμένα πράγματα για τις ε, τροπολογίες ε, που παρουσίασε η συγκήτρια. Κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε την εργασία σας και τη δική σας και των σκιωδών εισηγητών. Ε, νομίζω ότι η σύνοψή σας των τεσσάρων σημείων είναι πάρα πολύ σαφής και πολύ χρήσιμη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε γενικές γραμμές ε, έχει υποστηρίξει τις επίσημες στατιστικές και έχει τονίσει τη σημασία πιο συγκρίσιμων και πιο έγκαιρων στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι μια προτεραιότητα πολύ βασική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επίκαιρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, ε, αντικειμενική ε, ε, ενημέρωση. Ε, είμαστε σε πολύ μεγάλη πίεση για διάφορους λόγους ε, και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε σκοπό να, να αναμορφώσουμε πλήρως το πρόγραμμα. Θέλουμε, επεκτείνοντας το πρόγραμμα, να συνεχίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που έχει όλο και περισσότερες προκλήσεις να αντιμετωπίσει και να καλύψει πολλά αιτήματα ε, όταν γίνονται περικοπές στον προϋπολογισμό από τα κράτη-μέλη. Βλέποντας λοιπόν τα σημεία αυτά που έθεσε ε, η κυρία Αρένα, τα περιφερειακά ζητήματα, ε, το θέμα των ομάδων των ατόμων ε, με αναπηρίες, ε, ε, το θέμα της παραγωγικότητας και το συσχετισμό των δικτών. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ήδη επεξεργαζόμαστε, έχουν δρομολογηθεί, κάποια έχουν εξελιχθεί περισσότερο από άλλα. Όλα υπόκεινται στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε την νομική ε, βάση για να μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία των κρατών μελών για συνεχιστή παραγωγή των ποιοτικών στατιστικών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είδατε και στην πρόταση, εμείς έχουμε σκοπό να σημειώσουμε πρόοδο ειδικότερα σε φιλόδοξους τομείς, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε και τη μεθοδολογία και ε, τις δυνατότητες υπολογισμού που έχουμε. Εμείς ε, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και ε, με την εισηγήτρια, σε περισσότερες λεπτομέρειες και με την εισηγήτρια και ε, με την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ τη σύντομη παρέμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκερίκε, μήπως θέλετε να πείτε κάτι ως κοιόδης εισηγητής. Όχι. Καλώς. Να δώσω τότε το λόγο στην Μαρία Αρένα θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί των συμβιβαστικών τροπολογιών. Βεβαίως θα έρθουμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια καλή κατανόηση των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών που θα υποβληθούν και βεβαίως θα εργαστούμε για να καλύψουμε ε, τις ανησυχίες όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 13 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι έγκριση στις 22 Μαρτίου στην Επιτροπή μας ε, και ψηφοφορία στην Καθήλυνη Επιτροπή, Καθήλυνη Αρμόδια Επιτροπή στις 27 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της προβολής στις επιδόσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή και τον και αντιπρόεδρο Κλοντ Γούλαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το να ενισχύσουμε τη συνοχή και να προβάλλουμε τις επιδόσεις που θεωρώ ότι είναι βασική στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που συμβάλλουν επίσης στην εκπλήση των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη και αν ορισμένοι στόχοι ε, βρίσκονται σε καλή πορεία, άλλοι όπως η μείωση των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της στόχιας ε, απέχουν πολύ από την επιτεύξή τους. Η γνωμοδότηση αυτή προς την Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης αφορά δύο ζητήματα, την δέσμευση των εταίρων στην εκτέλεση των ταμείων, και η βελτίωση, τη βελτίωση της προβολής των ταμείων αυτών στους ε, πολίτες. Αυτό που μας ασχολεί, απασχολεί εμάς στην Επιτροπή μας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζω ιδιαίτερα, δίνω ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ταμείο φροντίζοντας ωστόσο η, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης να ε, αφορά και τα δύο θέματα. Υπερβολικά πολλοί πολίτες αγνοούν την ίδια την ύπαρξη των ταμείων αυτών. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, μόνο το 1 τρίτο έχει, τα έχει ακούσει και γνωρίζει ότι συγχρηματοδοτούνται τα λόγω προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Επίση, είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων επικοινωνία και να τα καλέσουμε να επιμείνουν στα θέματα, στην προστέμενη αξία σε θέματα απασχόληση χρειάζεται να επανεξετάσουμε τον κανονισμό 1303 του 2013 για να λεφθεί καλύτερα υπόψη η ιδιαίτερη φύση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να υπογραμμιστεί ε, μια συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκή για την οικοδόμηση ενός κτηρίου παρά για μια διαδικασία ένταξης ή ενσωμάτωσης. Για να έχουμε τη δέσμευση λοιπόν των εταίρων θα πρέπει να φροντίσουμε να μειωθεί το διοικητικό και οικονομικό άχθος ε, ε, στοιχεία που αποθαρρύνουν πολλούς φορείς ε, και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δυνατότητα τους να συμμετέχουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εμπνευστεί από την Τριμερή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς εταίρους, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα. Τέλος, παρότι είναι κάτι που υπάρχει, θα ήθελα τα κράτη-μέλη να αφοσιώσουν κάποιους πόρους του Ευρωπαϊκού Νομικού Ταμείου για την ενίσχυση των δημοσίων αρχών και τους κοινωνικούς εταίρους. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω τι συμμετοχέ των ΜΕΝ και των ΔΕ. Ευχαριστώ. Thank you. Then I give the floor Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Τζεντήλε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά την ε, εισαγωγική παρουσίαση αυτή της συζήτησής μας. Πρέπει να πω ότι ουσιαστικά συμφωνώ με τη δομή. Ε, είναι αναγκαίο οι πολίτες ε, της Ευρώπης να γνωρίζουν καλύτερα τις ευκαιρίες ε, που προωθεί η Ευρώπη στις διάφορες περιφέρειες αλλά και τα αποτελέσματα που αυτή η τεράστια προσπάθεια ε, επιτυγχάνει. Κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καλής ποιότητας. Και σίγουρα είναι θετική συμμετοχή ενδιαφερομένων ε, από το τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία μας λένε ακριβώς αυτό, ε, ότι τα ποσοστά που έχουν επιτυχθεί είναι ενδιαφέροντα όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μια εκτίμηση λοιπόν επιπτώσεων όσον αφορά την απασχόληση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό δίκτυ όχι μόνο όσον αφορά των πλέον εκτιμάτων ε, της πολιτικής συνοχής ε, αλλά και διότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο το οποίο θα αξιολογήσει την έκταση στην οποία η επικοινωνία, η ενημέρωση έχουν καταφέρει να ε, και να κινητοποιήσουν τους συνομιλητές μας στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Σίγουρα χρειάζεται και μια προσπάθεια μεγαλύτερης απλούστευσης ε, του κανονισμών, ε, της νομοθεσίας, γενικότερα της υποδομής και της αρχιτεκτονικής των διαρθρωτικών ταμείων. Σίγουρα υπογραμμίζοντας ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι έλεγχοι πρώτου και δευτέρου επίπεδου, ε, επιτυχάνουμε πολλά, αλλά κάτι που ακούμε διαρκώς σε συζητήσεις ε, σε διάφορες περιφέρειες είναι αυτό το αίτημα απλούστευσης. Από τη μία και της απλούστευσης της εκτέλεσης από θεσμική άποψη του δημόσιου τομέα που ε, εισέρχεται στην ε, εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, των ταμείων αυτών. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε κάποια προσοχή στις σχέσεις με τις αρχές των κρατών μελών όλα αυτά με το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εδώ θα ολοκληρώσω το όραμα αυτό το οποίο πρέπει να κοινοποιήσουμε περισσότερο, να ενημερώσουμε σχετικά με αυτό τους πολίτες, ειδικότερα τους πιο ευάλωτους, όσοι ε, απαιτούν να συμπεριληφθούν όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και πολύ συχνά οικονομικά από άψη εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προτάσεις μας ε, κινούνται προς αυτό που εμείς ευχόμαστε καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη γνώση, καλύτερη ενσωμάτωση, συντονισμό των ταμείων με μια δέσμευση ώστε να αξιοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενεργά στις πολιτικές ε, δημιουργίες της Ενεργασία. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, I will now... Ευχαριστώ. Κυρία Τρεμπέσιος, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συντάκνη γνωμοδότησης για την πάρα πολύ καλή του έκθεση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε. Ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία επανέρχονται συνεχώς είναι η ικανότητα των ε, εταίρων ε, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε τεχνική υποδομή και για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, αλλά και να δώσουμε χρηματοδότηση. Ένα από τα ζητήματα τα οποία καλύπτει η γνωμοδότηση είναι το διοικητικό άχθος. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, ε, όμως ε, η πρόκληση του να το κάνουμε αυτό χωρίς ε, να μειώσουμε τον απαραίτητο λογιστικό έλεγχο. Πρέπει εδώ λοιπόν να βρεθεί μια χρυσή Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, δεν διάβασα καλά το κείμενό μου. Θα ήθελα να πω πόσο σημαντική είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εξασφαλίσουμε ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο ε, ώστε να επιφέρουν προστιθέμενη αξία ε, επιπλέον της δουλειά των κρατών μελών. Για μας ε, υπάρχουν προτεραιότητες. Καταρχάς, η ενωσική χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδότηση εθνικών προσεγγίσεων, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επιπλέον υποστήριξη στους νέου κατά ώστε να ε, συμπληρώνεται και να ενισχύεται το εθνικό ε, πρόγραμμα κατόπιν απόφαση των κρατών μελών. Επίσης, ε, τα προγράμματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωση πρέπει να έχουν την απαραίτητη ευελιξία να ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν μια πιο μεμονωμένη προσέγγιση, ή να μπορούν να ε, προσανατολίζουν τη χρηματοδότηση στους τομείς και τις ε, περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερο τη χρηματοδότηση αυτή. Επίση, οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να βλέπει πέρα από το κόστος και τον αριθμό των ε, συμμετεχόντων και να βλέπουμε το κόστος σε πραγματικούς αριθμούς και να γίνεται σωστή ιεράρχηση όπως και κατανόηση του ε, πώς ε, και γιατί κάποιες δράσεις ε, είναι επιτυχημένες. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για να μπορέσω να να μπορέσει να, να καλυφθεί η άποψή μου στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Σελίμοβιτς. Ο κύριος Σελίμοβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την θετική του γνωμοδότηση. Είναι ε, μια βάση με την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε όλοι και να συνεργαστούμε μαζί του. Επειδή μόλι σήμερα έχω αναλάβει το έργο αυτό του σκιώδης εισηγητή, δεν θα προσπαθήσω να διατυπώσω πλήρω τι απόψεις μου. Θα επανέλθουμε όμως με τις ιδέες μας και τα κέρια σημεία εστίασης αργότερα με τις τροπολογίες μας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε κάποιες τροπολογίες σε κάποια σημεία τα οποία είναι προσφυλή σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε. Ευχαριστώ Ρίκη Πρόεδρος. Γκονσάλες Πένιας απουσιάζει. Κάνει άλλος δεν την εκπροσωπεί την ομάδα της ΓΚΟΕ. Πηγαίνουν στην ε, κυρία Ράνκε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και από τη δική μας πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία μοναχά τα οποία είναι σημαντικά αλλά δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Ένα είναι η δυνατότητα να δώσουμε την δυνατότητα συμμετοχής στην προετοιμασία των ε, σχεδίων και προγραμμάτων. Πολλές φορές η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να μην έχει την το μεγάλο, να μείνει το μεγαλύτερο μέρο τη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτονται από τοπικά και περιφερειακά κονδύλια για την προετοιμασία των σχεδίων ιδίως όταν πρέπει να, να υποστηρίξουμε μελέτες ή να κάνουμε λογιστικό έλεγχο για προγράμματα υποδομών. Εκεί υπάρχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είναι απαραίτητο αυτό να καλυφθεί περισσότερο, γιατί στο τέλος όταν έχει καλυφθεί το κόστος ενός σχεδίου από εθνικούς πόρους είναι πιο κοντά στην, είναι πιο ορατό και υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από ό,τι όταν έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκό ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε εμεί να μεταλαπαδέσουμε περισσότερο τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτών των σχεδίων. Και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι σημαντικό για την ομάδα μου είναι η έννοια τη εταιρικότητα. Δεν αναφέρεται εκπεφρασμένα. Όταν θέλουμε να συμμετάσχουν και οι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ και η κοινωνία των πολιτών σε ένα σχέδιο, αυτό είναι γιατί μπορούν να παίξουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για να κάνουν σαφέστερο το ότι υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ένα σχέδιο γιατί πολλές φορές δεν ε, είναι ορατό αυτό, είναι απαραίτητο λοιπόν όχι μόνο να έχουμε τις ταμπέλες που δείχνουν ότι έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να έχουμε τα δίκτυα ανθρώπων που μπορούν να τονίσουν και προς συμπολίτε τους το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες, αλλά αυτά ήθελα να πω για την έναρξη της συζήτησης και προσβλέπω στην συνεργασία με τον εισηγητή και τους αρσκιώδης. Ευχαριστούμε από το FDD. Λωράγια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Το Ταμείο Συνοχής είναι βασικό εργαλείο, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό που βλέπουμε στην πρόταση Omnibus. Πρέπει να βοηθά ε, να εξαλειφθούμε τις ανισότητες. Πρόκειται για πολιτικές που όπως και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να έχουν σημαντικά ε, αποτελέσματα για τα θέματα απασχόλησης και ποιότητα ζωής στον κόσμο, ειδικότερα στις περισσότερο μειονεκτούσες περιοχές. Για τη βελτίωση των επιδόσεων χρειάζεται συμμετοχή ευρεία όλων των μερών από το ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τους τοπικούς οργανισμούς με διακυβέρνηση προσεκτική και αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών που επιτρέπουν την πρόσβαση στα ταμεία και στις χρηματοδοτήσεις, χωρίς να μειωθεί η αυστηρότητα των ελέγχων. Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να καθορίζονται για κάποιο ε, χρονικό διάστημα μεγάλο και εκεί να συμμετέχουν άνθρωποι ικανείς χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κόσμος ε, βλέπει τα πράγματα λάθος λόγω των ε, όσων μαθαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, συχνά εστιάζονται ε, ειδήσει σε μεγάλα ποσά που φτάνουν, τα οποία δεν μεταφράζονται σε δημιουργία θέσεων εργασίας ή εστιάζονται σε υποθέσεις απάτης. Το κίνημα των πέντε θεωρεί ότι Κατά βάση πρέπει να ε, κοινοποιούνται οι διαγωνισμοί με κάθε μέσο, με τα κλασικά μέσα αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με, με ενημέρωση και κατάρτιση από, τους τοπικούς, ε, από αρχές για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Τα αποτελέσματα όπου υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να διαδίδονται, να αποτελούν το αντικείμενο ενημερώσεις, αλλά να κοινοποιούμε και αυτά που δεν λειτουργήσαν ώστε επικοδομητικά να διορθώνουμε τα λάθη για να βελτιωθεί στο μέλλον η εφαρμογή. Σε αυτά όλα βασίζονται οι τροπολογίες που θα υποβαλούμε εμείς στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, κύριε Ο κύριος Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εταίρων και το πόσο ορατή ε, είναι ε, στο πλαίσιο των επενδυτικών ταμείων και των διαρθρωτικών ταμείων, το σχέδιο γνωμοδότησης δεν μας φαίνεται ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Ο κύριος ε, Ρολά ε, λέει ότι είναι θλιβερό το γεγονός ε, ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συγχρηματοδότηση των έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι πρέπει όλες οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες. Ζητάτε περισσότερη ευρωπαϊκή προπαγάνδα για να δείξετε την προστιθέμενη αξία την ευρωπαϊκή όσον αφορά την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ε, λέτε ότι ε, από τη μία πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και περισσότερες υποχρεώσεις για τους δικαιούχους και από την άλλη λέτε ότι το διοικητικό άχθος ε, που θα βαρύνει τις αρχές και τους δικαιούχους πρέπει να μεωθεί ώστε να εξασφαλιστεί, και αυτό είναι λογικό, ένα καλύτερο ποσοστό αξιοποίησης των κονδυλίων. Υπάρχει όμως αυτό το παράδοξο. Ε, κύριε Ρολέ, συμπεριλαμβάνει παρόλα αυτά η έκθεσή σας και κάποια θετικά σημεία. Μας αρέσει το γεγονός ότι θέλετε το διοικητικό άχθος για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θέλετε να μειωθεί. Όμως ε, οι πραγματικές σας προθέσεις ε, είναι να αυξηθεί το επίπεδο της ευρωπαϊκής προπαγάνδας που θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή, πάρα πολύ καλή και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, και ότι ο σκοπός σας είναι να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής και η ποιότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως κύριε Ρολά, ξεχνάτε ή μάλλον παραλείπετε να εξηγήσετε ότι δεν είναι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά των ε, φορολογουμένων κάθε κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα όσων είναι καθαρών, ε, εισφο, καθαρής εισφορής όπως για παράδειγμα η Γαλλία 9 δις ε, ευρώ. Ε, οι Γάλλοι ουσιαστικά ε, παίρνουν πίσω αυτά που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ότι τα χρήματα πέφτουν από τον ουρανό όπως, όπως προσπαθείτε να υπονοήσετε. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σαλβάη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να απαντήσει τα, τις ερωτήσεις που στρέφονταν προς εσάς. Έχετε το λόγο. <laughs> Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι ο Μάτο Σαλβάη, είμαι από την, ε, το Τμήμα Επικοινωνιών ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όπως επίσης και τον κύριο Μπούντα για την έκθεσή του. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη, πάρα πολύ σημαντική και ευπρόσδεκτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί κάθε δράση που πηγαίνει προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης καλύτερης ενημέρωσης, περισσότερης διαφάνειας και μεγαλύτερης επικοινωνίας, Ω ε, ε, ως προς τα συγχρηματοδοτούμενα ε, έργα είναι ευπρόσδεκτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, επειδή υπάρχει κοινή διαχείριση, όχι μόνο το πρόγραμμα όχι μόνο η συνδιαχείριση δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα αλλά και την επικοινωνία. Είναι ένα διαφορετικό ε, στάδιο τη διαδικασία. Ξεκινά από τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνει στι εθνικέ τοπικέ περιφερειακέ αρχέ, και μετά φτάνει μέχρι τους δικαιούχους ε, του ε, project. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε το δίκτυο όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ως προς την κατανόηση του πώς δαπανώνται τα κονδύλια. Προσπαθούμε να το κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλουμε καταρχάς να ενισχύσουμε την συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης στα τοπικά. Είναι μία από τις ελάχιστες πολιτικές ε, που σημαίνει ότι ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους πολίτες ε, σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες. Κατά δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση που έχουμε με τη διαχειριστική αρχή, την τοπική αρχή, να υπάρχει μια κοινή πολιτική επικοινωνία και πηγαίνουμε προς ε, μία προσέγγιση που μοιάζει με εκστρατεία. Ε, πέρσι, για παράδειγμα, ζητούσαμε από τους δικαιούχους ε, να ανοιχθούν προς τους πολίτες, να δείξουν δηλαδή στους πολίτες τι ακριβώς κάνουν. Ε, είναι και η 60η επέτειος ε, ε, του, των διευθυντικών ταμείων και γι' αυτό προσπαθούμε με αυτήν την εκστρατεία να ευαισθητοποιήσουμε πολύ περισσότερο τον κόσμο και κάτι ακόμη που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε λίγο τον τόνο της επικοινωνίας μας γιατί μερικές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε πάρα πολύ θεσμικοί. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε κάπως πιο συναισθηματικοί, για να το πω έτσι. Ε, αυτό προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, βέβαια, πολλοί βουλευτές που πήραν το λόγο πριν από μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ε, η σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία ε, του αποτελέσματος της υλοποίησης ε, του έργου. Και τέλος, ε, επειδή λέτε ότι υπάρχει μία έρευνα που έγινε του Ευρωβαρομέτρου, θα υπάρχει μία ακόμη το Μάιο του 2017, σας το λέω αυτό για ενημερωτικούς λόγους, και θα μπορέσουμε πιο μετά να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Thank you for... Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόλα, εισηγητή. Έχετε σχόλια. Να ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συνομιλητές μας για τις διάφορες παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα για να καταλήξουμε σε σημαντικούς συμβιβασμούς, διότι άκουσα πολλά κοινά στοιχεία που μας απασχολούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η απασχόληση είναι κάτι που μας απασχολεί. Ε, πρέπει να επιμείνουμε στο πόσο ανάγκη είναι να αξιοποιήσουμε τις πολιτικές, να τις προβάλλουμε ε, και να εξετάσουμε τι επιπτώσεις έχουν. Το θέμα της απλούστευσης, χωρίς όμως να χαλαρώσουμε τους ελέγχους, τα δύο αυτά πρέπει να, υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Η προβολή της υπεραξίας ε, κυρίως των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα. Και τέλος, κάτι που μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι και μάλιστα δεν αναφέρεται ειδικότερα, ιδιαίτερα στο κείμενο που προτείνω, είναι ενισχυμένη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και οι συνεργασίες που θα πρέπει να υποστηρίξουμε, γιατί φυσικά οι συνεργασίες αποτελούν έναν πυρήνα ακρογωνιαίο λίθο ε, για την υλοποίηση αυτών των ικανοτήτων, αλλά και για την προβολή και την επικοινωνία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε καλή δουλειά για το μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρος. Η προθεσμία για τις είναι μέχρι τις 9 Μαρτίου. Έγκριση στην Επιτροπή Απασχόληση 2 και 3 Μαΐου και η ψηφοφορία στην ε, αρμόδια επί Επιτροπή 29 με 30 Μαΐου. Σας ευχαριστώ το σημείο 6 για τους ετούντες διεθνή προστασία αναβάλλεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και λόγω αυτού το απόγευμα μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο σημείο 8 της σημερινής διάταξης και είναι ευχής έργο ότι είσαστε παρούσα κυρία Σέβα που είστε η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια και την ε, Υγεία στον χώρο εργασίας, όσο ήρθατε στην Επιτροπή μας πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά δεν είχαμε τότε πολύ χρόνο στη διαθεσή μας και τρέχαμε για να προλάβουμε να τελειώσουμε τη μέση διάταξη. Τώρα είσαστε και πάλι παρούσα μεταξύ μας και μπορείτε να μας κάνετε μία παρουσίαση και σας δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν κυρία Σέντλατσεκ, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την... Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασιών του 2016. Τι κάναμε το τελευταίο έτος και θα σας παρουσιάσω και τα σημαντικότερα σημεία για την περίοδο του 2017 και 2018. Θα γνωρίζετε ότι η οσα συμβάλλει στην επίτευξη των κυρίων στόχων για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό. Τι εννοώ προκλήσεις ε, στα θέματα ασφάλειας στην απασχόληση. Αφορά τη γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη και την ανάγκη να διασφαλίσουμε ενεργό και υγιή γύρανση των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει ανάγκη συντονισμού των εθνικών στρατηγικών ασφαλείας και υγείας εστιαζόμενη στην υλοποίηση μετάφορα της σπουδαιότητα της χρήσης ε, συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Υπήρχε επίση πρόκληση διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό ασφαλείας, ε, ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίση αφορά το ε, πόσο σημαντικό είναι η σημαντική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασία, ώστε να διασφαλίζονται επαρκή επίπεδα πρόληψης ε, για τις ε, ασθένειες που σχετίζονται με το χώρο εργασία και την πρόβλεψή τους. Όλες αυτές οι προκλήσεις αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 ασφαλής και υγιής εργασία για όλους, εξυγχρονισμός ε, της σχετικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πολιτικών. Να αναλύσω τώρα τα όσα έγιναν το 2016. Πρώτον, είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον οργανισμό μας. Ήταν ένα έργο υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικία. Κάτι πολύ σημαντικό διότι αποτέλεσε τη βάση περαιτέρω συζητήσεων ε, και για την προετοιμασία της δικής μας εκστρατεία για τον υγιή χώρο για όλες τις ηλικίε ε, του 2016-2017 που τρέχει ακόμα. Στόχος του πιλωτικού έργου ήταν να προσθεθεί η υποστήριξη ε, στην βελτίωση των συνθηκών εργασία και στην ασφάλεια των εργαζομένων και εξάγαμε και κάποια συμπεράσματα για το τι αποτελεί καλή στρατηγική. Επίση, δώσαμε και κάποια παραδείγματα καλών στρατηγικών σε, σε επίπεδο επιχειρήσεων. Θα βρείτε τι πληροφορίε στην ιστοσελίδα μα. Υπάρχουν 29 εκθέσει χωρών όπου μπορείτε να δείτε ότι για 29 χώρες ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση του γυράσκοντος ανθρωπίνου δυναμικού. Και μετά παρουσιάζουμε μελέτες περιπτώσεων, προγράμματα στρατηγικές, ε, με ιδιαίτερη εστίαση στην αποκατάσταση, στην επιστροφή, στην εργασία. Και υπάρχει τώρα στην ιστοσελίδα μας και η τελική αναλυτική έκθεση που ενδιαφέρει όλους μας και ειδικότερα όσου είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής. αυτές τις δραστηριότητες είχαμε και τώρα έχουμε και τις δραστηριότητες αξιολόγησης ex post για να προσδιορίσουμε την προστιθέμενη αξία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την εκστρατεία του 2017 και 2018. Πρέπει να πω ότι συμμετείχαν όλα τα κράτη Μπέλη, η Νορβηγία, Ελβετία. Είναι σημαντική η πρόληψη σε όλο το χώρο εργασία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι εμεί δεν εστιάζουμε επαρκώ στου ε, πιο ηλικιωμένου εργαζόμενου και τα προβλήματά του. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε την πρόληψη ήδη όταν μπαίνουν στο χώρο εργασία σαν νέοι. Θα έχουμε λοιπόν την καταληκτική εκδήλωση σε αυτήν την ε, ε, εκστρατεία τον Νοέμβριο. Επίσης, ξέρετε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αξιόπιστα και ε, βασισμένα στην πραγματικότητα στατιστικά στοιχεία για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τους αναβιωμένους κινδύνους και είναι απαραίτητο να καλύψουμε το χάσμα αυτό πληροφορίες, να γίνουν έρευνες στις εταιρείε και με τον τρόπο αυτό να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας και της ασφάλειας σε επίπεδο ε, επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν δημοσίευσει και δευτερεύουσες αναλύσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και επίσης μια κοινή ανάλυση που κάναμε μαζί με την ε, έρευνα για, την, ε, για το ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο εργασίας για τα ατυχήματα και τις συνθήκες εργασίας. Συνεχίζουμε και άλλες ενέργειές μας για δευτερογενείς αναλύσεις, για τον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο και την επίπτωση του κινδύνου αυτού στο, στη διαχείριση των κινδύνων σε εταιρικό επίπεδο. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα που ξεκινήσαμε στο τέλος του 2015 μέχρι το 2016 ήταν για τους μετανάστες της επιχειρήσης. Ξέρετε ότι 93% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, για τις μικροεπιχειρήσεις, όχι για τους μετανάστες, για τις μικροεπιχειρήσεις έχουμε 93% μικροεπιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει την εκτίμησή μας για την κατάσταση το 2016 σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια για τις μικροεπιχειρήσεις. Συνεχίζεται λοιπόν αυτό το σχέδιο θα έχουμε τα τελικά μας πορίσματα το τέλος του 2017, αρχές του 2018 αν θέλει ο Γεραμπής και αυτό θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη και ποιοτικότερη ανάλυση των ε, σχημάτων συμπεριφοράς της μικροεπιχείρησης, για τον λόγο επίσης το ρόλο των ε, ενδιαμέσων και θα παρουσιάσουμε και πιο επιτυχή προγράμματα σε ένα διεθνές επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο. Επίσης έχουμε και μια διαδραστική, επιγραμμική αξιολόγηση κινδύνου και αυτό είναι από τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχολούν για τις μικροεπιχειρήσεις και αυτό είναι δωρεάν παρεχόμενο εργαλείο χωρίς κόστος και η Κομισιόν θεώρησε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί και η εμβέλεια αυτού του μέτρου και ζητά από τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν στα συστήματά τους το εργαλείο αυτό. Το 2016 λοιπόν, αλλά και το 2017, ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε με καλύτερο τρόπο το εργαλείο αυτό. Τι είναι αυτό το εργαλείο. Ήδη το 2016 <clears throat> έχουν υπάρξει κάπου 118 τέτοια εργαλεία, δύο το 2016 και άλλα 20 είναι εν ε, εξελίξη. Είναι σαν μια χιονοστιβάδα χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο γιατί συμμετέχουν όλο και περισσότερε εταιρείε. Το 2017 τώρα θέλω να αναφέρω ορισμένα προεξάχοντα στοιχεία γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας. Ο στόχος μας είναι να δούμε ποιοι είναι οι νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία που συνδέονται με τον αντίκτυπο των τεχνολογιών πληροφορίας και ε, υπολογισμών. Μιλάμε για τον ρόλο του υπολογιστικού νέφους ποιο ρόλο μπορούν να έχουν αυτά στο χώρο εργασία. Η μελέτη αυτή θα συμπληρωθεί το 2018 και έχουν ξεκινήσει και μελέτε σε σχέση με το μέλλον της εργασίας, κάτι το οποίο είναι ένα καυτό θέμα για όλους μας, γιατί ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει το 2017 είναι οι ασθένειες που έχουν να κάνουν με την εργασία και γυρίσουμε και στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των εργαζομένων οι οποίοι έχουν πληγεί από τον καρκίνο, επίσης ε, οι, αυτούς που έχουν θυγεί από έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες. Μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση της μεθοδολογίας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα αυτές τις ασθένειες με, την, ε, τον έλεγχο των ήδη υπαρχόντων συστημάτων εγγύρης προειδοποίησης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το έργο με επικίνδυνες ουσίες και αυτό θα αποτελέσει και τη βάση για την, μεγαλή, για την επερχόμενη επικείμενη μάλλον, εκστρατεία μας το 2018 2019 για τις επικίνδυνες ουσίες. Ένα άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει σίγουρα είναι η μακροχρόνια άδεια εργασίας λόγω ασθένειας και τα θέματα της προώρησης συνταξιοδότησης. Έχουμε ξεκινήσει ήδη μια γενική επισκόπηση. Έχουμε πολλά στοιχεία λοιπόν στον τομέα αυτό που μπορούμε να επεξεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των διαταραχών που μπορεί να έχει κανείς σε αυτές τις ε, περιπτώσεις για τις μειοσκελετικές διαταραχές συγκεκριμένα. Θέλουμε εκεί πέρα να εντοπίσουμε τα πιο σημαντικά εργαλεία παρέμβασης και να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα θέματα των μειοσκελετικό διαταραχών, αλλά τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη εστίαση γιατί το Διοικητικό μας ε, Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιανουάριο ότι αυτή θα είναι η εκστρατεία για τον υγιή χώρο εργασίας το 2020-2021 και εκεί λοιπόν θα εστιάσουμε στις μειοσκελετικές ε, διαταραχές μετά την εκστατεία για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων ουσιών. Τέλος, εμείς ε, λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματος 2014-2020. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει τώρα σε επίπεδο αξιολόγησης και ο, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας, αλλά συγχρόνως τον Ιούνιο θα αρχίσουμε να συζητούμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο τι θα μπορούσε να αποτελέσει τη στατική μας για το επέκεινα του 2020. Ξέρω ότι καταρχήν μου είχατε δώσει 10 λεπτά, εγώ πήρα μερικά περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες, για αυτή την ενημέρωση. Εμεί πρόκειται να συζητήσουμε τις αναθεωρήσεις για το ΙΟΣΑ αύριο το πρωί στην Επιτροπή. Αλλά και το κόσμο ακόμα ταξιδεύει, δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Αναφέρατε τους μεγαλύτερες ηλικία ε, τους γυράσκοντες εργαζομένους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν ερωτήσεις. Θα ήθελαν τα μέλη να κάνουν κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Σέτλατσεκ. Παρακαλώ κύριε Μπέκερ. Δεν είναι ερώτημα αλλά θα ήθελα να επενέσω αυτά που μας είπε η κυρία Σενέτσοβα, γιατί μπόρεσε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μας δώσει μια συνολική εικόνα και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία και σίγουρα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα από ό,τι μπόρεσε να πει και η κυρία Σενέτσοβα στο σύντομο αυτό διάστημα. Χακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι εισηγητής ε, για την εκθεσή αυτή και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Διευθύντρια, την κυρία Σέντλα για την παρουσίαση αυτή και για τις δραστηριότητες αυτές ε, που δίνουν πολλά στοιχεία και για τη δική μου έκθεση. και για τη συνεργασία του Συμβουλίου. Ήθελα να πω, κυρία Διευθύντρια, ότι ανοίγονται πολλές προοπτικές, πολλές προκλήσεις που αναλύσατε εσείς και που αφορούν την ασφάλεια ε, και την υγεία στο ε, χώρο εργασίας. Αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο το χώρο εργασίας στην Ευρώπη. Αναφέρατε την προστασία των νέων ε, που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, κάτι πολύ σημαντικό. Διότι είναι γυράς και ο εργαζόμενος πληθυσμός στην Ευρώπη, οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον των νέων. Διότι υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν επαρκή κίνητρα. Να θελήσει κανείς να μπει σε κάποιες δουλειές. Επίσης υπογραμμίσατε και κάτι άλλο σημαντικό, την επανένταξη στην χώρα εργασίας μετά από αποκατάσταση, μετά από θεραπεία. Πολλοί κόσμος ε, δυστυχώς ε, παραμένει απομονωμένος, αποκλεισμένος ε, μετά από κάποια ασθένεια. Αυτό δεν είναι σωστό οποιοδήποτε έχει περάσει από μια περίοδο σοβαρής ασθένειας και θεραπεία και αποκατάσταση θα πρέπει να, υπάρχει, να έχει πραγματικές δυνατότητες να επιστρέψει στην εργασία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο από ψυγεία και οικονομική άποψη αλλά και από κοινωνική άποψη. Δεν μπορούμε να ε, στιγματίζουμε τέτοιους ανθρώπους, να τους απομονώνουμε, να τους αποκλείουμε από την κοινωνία. Οπότε είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Και μετά εκεί όπου μιλάμε για την πρόληψη των νέων κινδύνων, ε, το να είμαστε προσεκτικοί, ε, να προβλέπουμε, να επιτηρούμε ε, και ογγλικά. Ο γιατρός πάντα λέει πρέπει να προσπαθούμε να προβλέπουμε, να κάνουμε ελέγχους. Ε, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι τα όσα λέτε είναι πολύ επικοδομητικά. Εγώ ως εισηγητής ε, θα έχω πολλά να πω φυσικά για το θέμα αυτό, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Ε, θα έχουμε και τις τροπολογίες. Ευχαριστώ την κυρία Διευθύντρια για την παρουσίαση. και που παρουσίασε τις διάφορες προκλήσεις με τρόπο ε, πολύ ε, συνεκτικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάχα. Ε, ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Σαντλατσέκ. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Αλλά αναφέρατε ότι βέβαια υπάρχει καθυστέρηση στο να έρθουμε στις Βρυξέλλες και έχουμε και πολλές επιτροπές. Δεν μπορούσα λοιπόν να ακούσω το σύνολο της παρουσίασής σας. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση για το πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ίση ε, προστασία για την υγεία και την ε, ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους με τις νέες μορφές που παίρνει η εργασία. Έχουμε, διατυπώσει, έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να έχουμε την ίδια προστασία σε μεγάλες και μικρές ε, επιχειρήσεις. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν την ασφάλεια και στις δύο περιπτώσεις. Και εσείς έχετε αναφερθεί και τις νέες μορφές, τις νέες μορφές εργασίας οι οποίες ε, αναδύονται. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς ως κοινωνία να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε προβλήματα υγείας και ασφάλειας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει εμείς να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Χάρκιν. Σας ευχαριστώ. Και θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για όλα αυτά που μας είπατε. Ε, όλα αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Κάτι που θα ήθελα όμως να πω είναι όταν ε, βλέπω το κομμάτι που αφορά τις ε, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πριν από λίγα λεπτά στη συζήτησή μας μιλούσαμε για τη μείωση του διοικητικού άχθους και πολλές φορές στο Κοινοβούλιο έχουμε την τάση, με τις καλύτερες των προθέσεων βεβαίως, να προσθέτουμε διοικητικό άχθος και είναι πολύ καλό να ακούμε από τη δική σας τη δουλειά ε, όσον αφορά τα ε, διαδραστικά ε, διαδικτυακά μεργαλεία ότι προσπαθείτε να μειώσετε το διοικητικό άχθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα στον τομέα των νέων αναδυόμενων κινδύνων, να κάνουμε μία προσπάθεια. Εμείς είχαμε πολλές εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ως Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά όσον αφορά τις μειοσκελετικές ε, διαταραχές ε, την ε, προηγούμενη θητεία εγώ ήμουν η συγγήτρια για μία πρόταση που αναμενόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τελικά δεν προχώρησε οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να πιέσετε για περισσότερη νομοθεσία στον τομέα αυτό. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Καταρχάς αναφερθήκατε στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ποια ε, είναι η εργασία σας ε, ή τι προγραμματίζετε να κάνετε ως προς ε, τον τομέα αυτό. Όσον αφορά τώρα την όλη ιδέα των συνεργειών των διαφόρων υπηρεσιών. Από τη δική σας προοπτική πώς προχωρά αυτή η προσπάθεια και επίση ε, η εκστρατεία για τους ασφαλέστερους χώρου εργασίας. Πάρα πολύ σημαντική η δουλειά σα. 29 χώρε μελετήσατε, υπήρξαν συγκεκριμένα παραδείγματα και δώσατε και παραδείγματα ε, του πώ ε, διοχετεύονται οι πρακτικές. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε ε, πώς κάνατε την ανάλυση ε, των αποτελεσμάτων ε, ή τον υπολογισμό των διαφόρων στοιχείων σας. Και θα ήθελα επίσης να επανεπισημάνω αυτό που υπόθηκε για τις νέες μορφές εργασίας, μιλήσατε για τη συνεργατική οικονομία, εμείς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Έχετε σχέδιο έχετε προγραμματίσει να δείτε κατά πόσο και πώς επηρεάζει αυτό τους εργαζόμενους, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο τελικά πλησιάζει με αλματώδη βήματα και θα θέλαμε να μπορέσουμε να ε, δούμε την ενδεχόμενη νομοθεσία, ε, τη ρύθμιση που χρειάζεται και χρειαζόμαστε και πολύ καλή ενημέρωση για να το επιτύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δίνω το λόγο στην κυρία ε, Σέντλατσο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς ε, γιατί επενέσατε τόσο πολύ τη δουλειά μας. Ε, κύριε Χόκ, όταν αναφέρατε την σημασία της συμμετοχής των νέων και των γυρεότερων εργαζομένων ε, η ανάλυση μας ε, των δραστηριοτήτων μας και των προγραμμάτων μας έδειξε ότι χώρες κυρίως που έχουν μία ε, πιο σφαιρική προσέγγιση για τη διαχείριση του γυράσκοντος εργατικού δυναμικού ε, είναι οι χώρες οι οποίες ε, έχουν σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία και επίσης ε, έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό νέων και γυρεότερων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν το ευρύτερο πρόγραμμα που έχει αυτή τη σφαιρική προσέγγιση ε, αφορά τέσσερις ομάδες χωρών και η μία ομάδα, η πρώτη, είναι αυτή που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Η αποκατάσταση από προβλήματα υγείας είναι ένας πολύ βασικός τομέας και εδώ βλέπουμε μεγάλη επιτυχία με την συμμετοχή υγιών ανθρώπων που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εργασία τους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά συμπεράσματα που μπορέσαμε να εξαγάγουμε από ε, την ανάλυση αυτή. Όσον αφορά τώρα και θα μιλήσω γερμανικά τώρα. Ποιος μου έκανε αυτή την ερώτηση. Νέες μορφές ε, συμβάσεων εργασίας. Ε, αλλάζει ο κόσμος της εργασίας και αλλάζουν και οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και επανήλων. Και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον. Στα προγράμματά μας για τα ICT και τους χώρους εργασίας ε, που διαφέρουν από τους παραδοσιακούς. Πιθανότατα τέλη του έτους, εντός αυτών των προγραμμάτων, θα διοργανώσουμε κάποια διάσκεψη ή κάποιο σεμινάριο και με την ευκαιρία αυτή ελπίζουμε θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε τα πολιτικά επίπεδα, για παράδειγμα να προσκαλέσουμε υπουργού απασχόλησης, οι οποίοι ήδη έχουν εισάγει κάποιες αλλαγές στην ομοθεσία τους. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε τον κύριο Γιονκέρο, ο οποίος ανέφερε κάποια πράγματα για τον κοινωνικό πυλώνα, είχαμε συζητήσει με του υπουργού από τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Γερμανία και ορισμένους άλλους, οι οποίοι ήδη στην νομοθεσία τους έχουν νομοθετήσει ήδη για αυτές τις νέε μορφέ εργασία. Εγώ ως Αυστριακή το γνωρίζω και ξέρω ότι γίνονται πολύ καλές συζητήσεις για το πώς θα καθορίσουμε τι σημαίνει απασχολούμενο σε σχέση με την παραδοσιακή έννοια. Ε, σε ε, το μίσο όπως το cloud computing για παράδειγμα. Οπότε θέλουμε να κάνουμε μια έκκληση να συζητηθεί σε τι σημαίνουν όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο και πώς μεταφράζονται σε νομοθεσία ώστε να υπάρχει μια γρήγορη αντίδραση. Πάω πίσω, περνάω πίσω στα αγγλικά. Ε, yes, ε, what we do is... Λοιπόν, τι κάνουμε. Σε αιτήσια βάση Θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση με τις ε, οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τη Eurofound, Sendefop και άλλους. Και ειδικότερα με τη Eurofound, ε, κάθε χρόνο υπογράφουμε μια συμφωνία μεταξύ της EOSA και της Eurofound, όπου συμφωνούμε να συνεργαστούμε επί συγκεκριμένων τομέων. Επίσης, ε, εκπονούμε και μια δημοσίευση ε, έχουμε και μια δημοσίευση για τη γύρανση του, των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά φροντίζουμε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Είναι σημαντικό να συμφωνούμε επί των προγραμμάτων εργασίας, επί συγκεκριμένων θεμάτων και πιστεύω ότι Όλοι μας ε, θέλουμε να θέσουμε στόχο να μην έχουμε επικαλύψεις, παρότι φυσικά αυτό είναι ένα απόφευκτο φορέ. φορές. Επίσης ρωτήσατε για την εκστρατεία για την υγεία στο χώρο εργασίας και πώς επηρεάζει η εκστρατεία υγείου χώρου εργασίας στο ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. Εμείς ε, πραγματοποιήσαμε και μόλις ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση της προηγούμενης εκστρατείας ε, υγιούς χώρου εργασία για τους ψυχοκοινωνικού κινδύνους και μόλις είδαμε την έκθεση, ε, μόλις ε, έφτασε και σε μένα και από την πρώτη ανάγνωση ε, έχω σχηματίσει θετικέ εντυπώσεις. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά κάνουμε το ίδιο για όλες αυτές τις εκστρατείες. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι ότι φυσικά είναι σημαντικό σε εθνικό επίπεδο ε, τα εθνικά μας δίκτυα ασφάλειας και υγείας ε, να εμπλέκονται, να συμμετέχουν, να ε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Αυτή δεν πάει να είναι ακόμα και σήμερα μια από τις συστάσεις παρακαλούμε στο εθνικό επίπεδο να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο δραστήρια εμεί θα εξελογήσουμε όλε τι εκστρατείε για την υγεία στον χώρο εργασία και πρέπει να πω ότι αποκτάμε όλο και περισσότερε επιχειρήσει ω εταίρου, όλο και περισσότερου εταίρου γενικότερα. Αλλά φυσικά πάντα υπάρχει χώρο περιθώριο βελτίωση ε, και να προσθέσουμε και άλλα μέλη τα οποία θα συνεργαστούν μαζί μα. Το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν κατάλαβα πολύ καλά, να σα πω την αλήθεια. Ρωτήσατε αν είναι τομέα που μας απασχολεί, αν έχουμε δραστηριότητες, αν έχουμε προγράμματα. Ναι, διάβαζα την παρουσίασή σας και έλεγε ότι το 2017 θα φέρει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μίλησε για τον Ευρωπαϊκό Πλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και κάποια από αυτά ενισχύουν τη σπουδαιότητα του έργου της EU όσα κτλ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το κύριο μας θέμα είναι η ασφάλεια και η υγεία. Για μας είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το να έχουμε μια, ένα χώρο εργασίας όπου ισχύει η υγεία και η ασφάλεια. Και ιδίω το σχέδιό μας για την γυράσκον δύναμη εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση και στον κοινωνικό τομέα που έχει επιπτώσεις στην κατάσταση ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως κομβικά και στο επίκεντρο το θέμα της υγείας και ασφάλειας και αυτό θέλουμε να έχουμε μια δύναμη εργατική η οποία είναι ασφαλής και υγιής. Uh, Ελπίζω ότι έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματά σας. Ναι, ναι, και εγώ πιστεύω ότι το πράξατε, λέει η κυρία Ουλσκοκ. Επομένω, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, όχι σήμερα φυσικά. Θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Θα, θα συζητήσουμε προηγουμένω τα ζητήματα αυτά για τα ζητήματα της ΩΣΑ και του ΣΕΔΕΦΟΠ. Μα θα θέλαμε λοιπόν επομένως να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Πάντοτε είσαστε καλόδεκτοι και τα θέματα αυτά αποτελούν και τις ε, κομικές αξίες της Επιτροπής μας και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε το ταχύτερο δυνατό και τούτου λεχθέντος. Έχει τελειώσει η συνεδρίασή μας, αλλά μην το ξεχάσετε 9 το πρωί έχουμε να ψηφίσουμε. Ελάτε λοιπόν να μην ξεχαστείτε. Ευχαριστώ. Thank you for the